So the first one is without voting list. It's just by show hands. Okay. Okay. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Προεδρεύουσα κυρία Χίρς, ας αρχίσουμε τώρα και να προχωρήσουμε γρήγορα. Θα αρχίσουμε με την πρώτη ψηφοφορία, το υπαριθμό 25 δηλαδή, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Έχουμε μια επιστολή να ψηφίσουμε την οποία γνωρίζετε. Παρακαλώ να γίνει ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή ηλεκτρονικά, αρχίζει. Τέλος. 40 υπέρ, μία κατά. Εγκρίνεται επομένω. Το υπαριθμόν 26. Αρμοδιότητες του, κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή οδηγίας του Συμβουλίου κτλ. Η συμφωνία που συνήψαν οι Ένωση Ευρωπριστών και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές σχετικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006. Τώρα, ψηφίζουμε για την Συμφωνία Πρώτης Αναγνώσεως με το Συμβούλιο. Αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Τέλος. 40 υπέρ, μία ψήφος κατά και επομένως εγκρίνεται. Ακολουθεί έκθεση για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης, η έκθεση της κυρίας Κίνγκα Γκönς. Συμβαστική Τροπολογία υπαριθμών α. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία L. Όπως λάμδα διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. ακολουθεί η τροπολογία 9 της κ. Ζούμπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οι υπαριθμούν 10 πάλι του ίδιου όνομα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή συμβαστική β λαϊκό κόμμα σοσιαλιστές δημοκράτες φιλελεύθεροι και πράσινοι ψήφι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική ΙΑ. Ίδιες πολιτικές ομάδες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΙ. Πάλι ίδιες πολιτικές ομάδες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Ζούμπερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική G. Ίδιες πολιτικές ομάδες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική σε γάμα. Πάλι ίδιες πολιτικές ομάδες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F πάλι των ίδιων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική D δέλτα υπέρ, υπέρ κατά από, όχι, αποχές τώρα μάλιστα εγκρίνεται. Τροπολογία 40 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή. Συμβαστική ε Λαϊκού Κόμματος Ασυμικρατών ναι, ναι, ναι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική HB ή τα Β των ίδιων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμών 53 της κυρίας Γκένς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική Age με τις ίδιες πολιτικές ομάδες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Age A. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομοίως. 62 Μπέκερ. Αυτή όμως έχει μόνο γλωσσικό χαρακτήρα και δεν ψηφίζεται επομένως. Ακολουθεί η υπαριθμόν 68 του κυρίου Μπεναμιάς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 Βαντερστούπ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική J των ίδιων πάντα πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική IB, ΙΒ, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική K, πάντα οι ίδιες πολιτικές ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 97 της κυρίας Κρόνς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 Βαντερστούπ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία που γίνεται ηλεκτρονικά Πέρας. 38 υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές. Εγκρίνεται επομένως. Συγχαρητήρια κυρία Συγγήτρια. Um, 27. No. 28. So. next on the agenda is... Ακολουθεί τώρα ο προπολογισμό 2014. Εντολή για τριμερή διάλογο με εισηγητή τον κύριο Σάβα Όρη. There problem? No, no, no. Okay. Good. Then we can start with the votes. Ας αρχίσουμε τότε. Πρώτη τροπολογία του κυρίου Νταρντέν υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α. Επιπλή Αλτε πράσινη. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 Νταρντέν. Με προφορική τροπολογία Υπάρχουν μήπως ενστάσεις, όχι, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τέλος, πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας είπα. 18 υπέρ και 23 κατά. Απορρίπτεται. Η 6 της κυρίας Γκόνς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 7 Ζούμπερ υπέρ κατά απο... αποχές απορρίπτεται. 8 πάλι Ζούμπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 πάντα της κυρίας Ζούμπερ υπέρ Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Συμβαστική Β. Λαϊκό κόμμα, σοσιαλδημοκράτες, άλλοτε και πράσινοι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπαριθμόν 12 ζούμπερ, υπέρ, κατά, αποχές, από 13 των κυρίων Νταρντέν Γκέν Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 ζούμπερ υπέρ κατά αποχές αυτή απορρίπτεται 15 Νταρντέν Guns υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 Λάμπερτ υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 17. δεν. Εδώ προβλέπεται κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα χωρίς το κείμενο ζητεί από την Επιτροπή κλπ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και αυτό. Νο, όχι με συγχωρείτε, απορρίπτεται, με συγχωρείτε. 18 μπουλόν. Αυτή είναι συμβατή με την υπαριθμό 17, αλλά την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική σι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 Δαρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 της κυρίας Ζούμπερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ε, λαϊκού κόμματος και λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33, Νταρντέν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία τώρα αρχίζει αφού θα γίνει ηλεκτρονικά. Πέρας. 36 υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Άρα εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Um, Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Κοσλόφσκι για τις συνέπειες των δημοσιονομικών περιορισμών για τις τοπικές αρχές όσο αφορά τα πάνε των διαρθρωτικών ταμείων. Συμβιβασμός Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 McIntyre, ε, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, χωρίς τη λέξη less, υπέρ, υπέρ του πρώτου τμήματος της 5, κατά, αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 23 υπέρ 16 κατά 3 αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Με τη λέξη λες. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός Β. και σοσιαλιστές και άλλοι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 McIntyre υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται ε, συμβασμός CL και σοσιαλιστές φιλελεύθεροι και άλλοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 Κοτσολίνο ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα με προφορική τροπολογία τονίζει επιπλέον ότι από το συνολικό ποσό των 11,2 δις που προβλέπονται στον ε, διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 2 κάθετος 13, 3.225 ε, δις ορίζονται για το ΕΚΤ που θα πρέπει να καταβληθούν σε δύο τμήματα. Αντιτίθεται κάποιος, φαίνεται πως όχι, ξεχωριστή ψηφοφορία που ζήτησε το ΕΛΚ, άρα καταπίπτει, τη στιγμή που εγκρίνουμε την προφορική. Δεκατρία όπως έχει τροποποιηθεί με την προφορική. Με τη λέξη bear. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Δεν πρέπει, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα, γιατί η λέξη δεν ε, υπάρχει στο κείμενο. D, ΕΛΚ, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι, πράσινοι, ευρωπαίοι ε, μεταρρυθμιστές και συντηρητικοί. Okay. We have the word bear has been taken out. Yeah. No, we don't have to vote on the second. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα, διότι η προφορική άλλαξε το πρώτο τμήμα και επειδή την εγκρίναμε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Εντάξει, καταλάβατε. Δέλτα. ΕΛΚ, σοσιαλιστές, ε, φιλελεύθεροι κλπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται ε, ΕΛΚ, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17, κοτσολίνο. Α, με συγχωρείτε, πίπτη, 21, Μακεντάιερ, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 21. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ 18 κατά. 22 Σρέτερ ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα χωρίς τη λέξη particularly υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε αρχίζει η ψηφοφορία ελέγχουμε Πέρας. Απορρίπτεται με 23 ψήφους κατά και 16 υπέρ. 23 Σρέτερ πρώτο τμήμα, χωριστή ψηφοφορία, τονίζει τον ρόλο μέχρι το job creation υπέρ. Κατά αποχές απορρίπ... εγκρίνεται, με συγχωρείτε. Δεύτερο τμήμα, αποκαθιστώντας την κινητικότητα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε ελέγχουμε ηλεκτρονικά Vote is closed. Πέρας. 23 υπέρ, 19 κατά, άρα εγκρίνεται. Τροπολογία 24 της κυρίας Σρέτερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 μπένιον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 Εσάια υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά πέρας 22 υπέρ 21 κατά άρα εγκρίνεται Συμβιβασμός G, L, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι, Πέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31, Εσάια, προφορική. Τροπολογία της κυρίας Εσάια. Ε, μιλάμε για τη χρήση κονδυλίων και μετά γίνεται η διαγραφή έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθ' τη διάρκεια, την, ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει το Embedded Communications Leading. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32. στουπ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός HL και σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι και άλλοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 Νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 καταπίπτει Άρα ε, αρχίζει η ψηφοφορία επί του τελικού κειμένου. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 43 υπέρ, ένας κατά, καμία αποχή. Να, συγχα... να σας συγχαρούμε, ενεκρίθη η έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Deutsch πρόσβαση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών της Ένωσης στην αγορά τρίτων χωρών στο μέτρο των δημοσίων συμβάσεων. Αρχίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 22 Σίπελ και ΚΑΣΤΕΞΕ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, από το ΕΛ και σοσιαλιστές υπάρχει ένας υπεράριθμος από το, στους, ε, από το ΕΛΚΑ κόμμα. Υπάρχει ένας υπεράριθμος. Εντάξει τώρα. Πέρας. 24 κατάρα απορρίπτεται, έναντι 19, τροπολογία 23, Χέντελ υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. ΑΛΦΑ, συμβιβασμός υπέρ Θέλετε να ελέγξουμε την 23. Ωραία, ελέγχουμε την 23 ηλεκτρονικά. Vote is closed. Πέρας. Άρα εγκρίνεται 23. B, A, C, A, D. All these compromises are voted on block. Okay. Um, the next we... Λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε την α, α, α, β, a, c, a, d, a, e, a, g, a, f και α. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε αν μπλοκ της ε, τροπολογίας συμβιβασμού. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Άρα οι τροπολογίες συμβιβασμού εγκρίνονται. Και περνάμε τώρα στην 25. Σίπελ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 Νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος Β, ΕΛΚ και Σοσιαλιστές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός ΣΥ, και Σοσιαλιστές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δέλτα, ε, ΕΛΚ, Σοσιαλιστές Γκουίπερ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32, Χέντελ υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33, Χέντελ υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5, του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται 6 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 Σίπελ και Νταρντέν ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα το κείμενο χωρίς ε, τις λέξεις but shall be rather και labor situation υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 σίπελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 40. Πέρας. 24 κατά έναντι 19, άρα απορρίπτεται. 7. Σίπελ Καστέξ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Χέντελ υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Αρχίζει ο έλεγχος. Πέρας. 21 υπέρ, κατά 23, άρα απορρίπτεται. 10 σίπελ και καστέξ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 Σίπελ και Καστές, ε, Καστέξ ξεχωριστή η ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, όλο το κείμενο χωρίς λέξεις και που δεν τηρούν ε, σύμφωνα με την οδηγία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται με 26 υπέρ και κατά 18. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα. Καταπίπτει γιατί 11 είναι κρίφη, 12 χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 σίπελ και νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες από την 17 ε, έως την 21. Όχι. Ωραία, ξεχωριστά. Τροπολογία 17. Σίπελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Σίπελ Νταρντέν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Σίπελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 σίπελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 σίπελ και νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 34 υπέρ, 7 κατά, 3 αποχές. Να συγχαρούμε την ε, εισηγήτρια. Το επόμενο θέμα είναι ο κανονισμός για τα ηλεκτροτεχνολογικά προϊόντα για τροποποίηση οδηγίας 2001-83 και του κανονισμού 178-2002 και 1223-2009. Η κυρία Στρέλα είναι η εισηγήτρια. Αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Με την 28 και 29 που είναι παρόμοιες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 23 υπέρ, 18 κατά, άρα εγκρίνεται. 13 μπιτζότο υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε ελέγχουμε ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας. 23 υπέρ και κατά 20. Άρα η 30 εγκρίνεται. Euh, Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. 32 euh, και 34 είναι παρόμοιες, τις ψηφίζουμε από κοινού υπέρ, κατά αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 27 υπέρ 14 κατά 3 αποχές, άρα εγκρίνεται. 35 ε, παράγραφος 4 ε, υπέρ της διαγραφής κατά αποχές εγκρίνεται. Η 33 την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 Χάρκιν για διαγραφή υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε για την 36. Ψηφίσατε όλοι πέρας 25 υπέρ 17 κατά άρα εγκρίνεται 37 η 37 έχει αποσύρθει και τώρα ψηφίζουμε την 4 ε, διότι 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 έχουν αποσύρθει 4 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51. βιτζότο Για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 44, παράγραφος 6, συμβασμός σε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 πιτζότο για διαγραφή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 54 χάρκιν υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά σε παληθεύσουμε καλύτερα. Υπεράριθμη η του ΕΛΚ κατά 2. Εντάξει, καλύτερα τώρα. Πέρας. 27 υπέρ, 13 κατά. Άρα εγκρίνεται 55 Jean Lambert υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 56 του ιδίου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 57 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 9 της εισηγήτριας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 10 της εισηγήτριας για διαγραφή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 59 μπουλών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 60 χάρκιν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 11 της εισηγήτριας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 της εισηγήτριας με μια προφορική των φιλελευθέρων. Κανείς δεν αντιτίθεται, άρα ψηφίζουμε την 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 της εισηγήτριας σε δύο τμήματα, το πρώτο τμήμα χωρίς τη λέξη and review μέχρι professional organization υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της προσθήκης των λέξεων υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα. Ελέγχουμε. Il y a un υπεράριθμο το ΕΛΚ κατά έναν. Εντάξει, ψηφίσατε όλοι. Nous votons la deuxième... Ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 14 και η συγγήτρια είναι υπέρ. Bien. J'ai l'impression que les choses se sont clarifiées. Le Πέρας. 38 υπέρ. 6 κατά. Με μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται. Στο, στην αιτιολογική σκέψη 2 ε, α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 Τροπολογία 16. Μπουλό με μια προφορική των φιλελευθέρων. Κανείς δεν αντιτίθεται. Γι' αυτό ψηφίζουμε τη 16 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 13, ε, τροπολογία 17 μπουλών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 έχει αποσυρθεί Άρα ψηφίσουμε 19 Φιλίπ Μπουλόν υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 20 ε, του ιδίου υπέρ. Κατά. Θα υπαλληθεύσουμε. Ελέγχουμε την 20. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 26 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. 21 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 του ιδίου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Β τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ε, υπεράριθμοι η του ΕΛΚ. Έχουμε έναν υπεράριθμο, τώρα εντάξει, 43 υπέρ, ένας κατά, καμία αποχή, να συγχαρούμε την εισηγητριά μας, την κυρία Στρέλα, η οποία απουσιάζει. Θα διαβιβάσουμε τα συγχαρητήρια. Να ψηφίσουμε εκ νέου έκθεση της συναδέλφου Στρέλα. Πρόκειται για την πρόταση κανονισμού για τα διαγνωστικά ιατροφημιλικά προϊόντα in vitro. Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1, τροπολογία 16, μπουλόν, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 39 παραγραφός 4, συλλογικό τμήμα, τροπολογία 3 της εισηγήτριας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 17 Κάρνουχ είναι συμβατή, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 42, παράγραφο 6, τροπολογία 4, τη εισηγήτριας, υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 18, είναι συμβατή, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, τη εισηγήτριας, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 6, τη ιδία υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Άρθρο 61, παράγραφος 1 από παράγραφος 1, τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 19 κάρπνο, έχουν συμβατή, ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Για το παραρτήμα 1, τμήμα 3, τροπολογία 8 της εισηγητρίας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Για το σημείο 17 τώρα πάλι του παραρτήματος 1, τροπολογία 20, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το εκτιμώντας α, συμβαστική πρόταση α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας 3, τροπολογία 10, μπουλόν, με προφορική τροπολογία από τους φιλελεύθερους, δεν υπάρχει αντίρρηση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας 13, τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το δούμε για το 11. Ψήφισατε όλοι, πέρας. 23 ψήφι υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. 12 του ιδίου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 του ιδίου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 του ιδίου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 του ιδίου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 Δύο της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά, αρχίδη ψηφορία. Ψήφισατε όλοι, πέρας. 44 υπέρ, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην συγγήτρια. Και τους κοιόδες βεβαίως. Φτάνουμε στο σημείο 33, στη γνωμοδότηση για την έκθεση πρωτοβουλία. Επιτροπή ε, ΙΜΚΟ, εσωτερική αγορά υπηρεσιών, περιγραφή της κατάστασης και επόμενα βήματα. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση του κυρίου Κάσα. Τροπολογία 1, Μέρφυ, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 του συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 τέλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόβος 1 τροπολογία 4 ζουμπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 μέρφη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά τα 1, τροπολογία 6, Καρυμαντέλη, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, της ιδίας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός α, από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά φτάνουμε στην τροπολογία 14, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 καρυμαντέλη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 της ιδίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 της ιδίας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 ζούμπερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 πολυμέρφη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 20 μαντέλι Πέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 21 αποσύρεται ψηφίζουμε λοιπόν την 22 της Γιούτα Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 Ζούμπερ Πέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 24 Γιούτα και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 έχουμε και προφορική τροπολογία εδώ δεν υπάρχει αντίρρηση επομένως ποιος είναι υπέρ έτσι όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά πάμε στην παράγραφο 3 τροπολογία 26 Κοτσολίνο με προφορική τροπολογία από το ΕΛΚ δεν υπάρχει αντίρρηση Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 27 είναι σούπερ, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεσμός Β από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 31, Μαρία Χάρκιν, για τμηματική ψηφοφορία το πρώτο τμήμα χωρίς ε, τις λέξεις in particular occupation all passion schemes υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 32 πολμέρφη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 του ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33, 34 συγγνώμη χείρση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 Γιούτα Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 Ντεβιτ Κάσε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε το συνολισμό της τη ψηφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 41 ψήφι υπέρ, τέσσερις κατά, καμία εποχή. Ωραία, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Non, Φτάνουμε στο σημείο 34 για να ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Για την προφορική ερώτηση. Έχουμε δύο τροπολογίες. Πρώτη τροπολογία παρουσιάστηκε από τον Αλχάντρα Σέρκος από τους σοσιαλιστές. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, έχουμε την εισαγωγή ενό νέου θέματος με τροπολογία 2 από τον κύριο Σέρκας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το συνολικό του ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 42 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Επομένως, εγκρίνεται η προφορική ερώτηση. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος, αυτή καθ' αυτή, ξεκινάμε μετακτημώντας. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να τα δούμε όλα μαζί. Μετακτημώντας β, σας προτείνω τροπολογία 1 του κυρίου Σέρκα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 που έχει αποσυρθεί και κατόπιν να ψηφίσουμε τροπολογία 3, Πατρικ Λεγιαρίκ και την ομάδα Γκου υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 1. Ψηφίζουμε το συμβασμό Α από δύο ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 2 έχουμε ένα τεχνικό λάθος, δεν πρέπει να το ψηφίσουμε λοιπόν αυτό. Το 2014 θα αντικατασταθεί με το 2013 και Και, ψηφίζουμε την τροπολογία 7. Το Αλεχάνδρο Σέρκα υπέρ. Κατά αποχέ συγκρίνεται τροπολογία 8. Πατρακλή συμβατή. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 9 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται ψηφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Λοιπόν, καλώ όλε τι ομάδε που ψήφισαν και υποστήριξαν αυτή την προφορική ερώτηση και την πρόταση ψηφίσματο να ασκήσουν πίεση στις ομάδες τους έτσι ώστε να μπορεί να γραφεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη τη Συνόδου του Ιουλίου. Γιατί διαφορετικά θα καθυστερήσουμε υπερβολικά. Φτάνουμε στο σημείο 35 για να ψηφίσουμε την έκθεση της Επιτροπής μας για την πρόταση οδηγία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 9671 σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων για τον κατάλογο των ψηφοφοριών έτσι όπως καταρτίστηκε ως πρόεδρος έπρεπε να καθορίσω τη σειρά των ψηφοφοριών, των τροπολογιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες πρακτικές στο Κοινοβούλιο και των αρμοδιοτήτων έτσι όπως έχουν καθοριστεί από τον εσωτερικό μας κανονισμό. Για το άρθρο 161, βάση του άρθρου 161, το θέμα της ψηφοφορίας, της σειράς των ψηφοφοριών τροπολογιών, άπτεται μια συζήτηση που βασίζεται ε, στον απομακρυσμένο μη χαρακτήρα του κειμένου σε σχέση με την αρχική πρόταση. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την προτεραιότητα, τότε λέει το άρθρο 161 ότι η πρόεδρος αποφασίζει. Αυτό το ξεκαθάρισα και από τον αρμόδιο γραμματέα που, είναι, που έχει αναλάβει το φάκελο. Επειδή είναι λεπτός ο φάκελος αυτό, ξέρω ότι οποιαδήποτε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση θα προκαλέσει συζητήσεις. Αλλά σας προτείνω να δεχτείτε την πραγματικότητα όσων έχουν αποφασιστεί. Έτσι λοιπόν ως ε, υπάλληλο αυτού του οίκου εγώ μπορέσα να λάβω αυτές τις αποφάσεις. Περνάμε στο συμβιβασμό ΒΒ2 άρθρο 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Παρακαλώ κύριε Συγήτρια, ναι, για το θέμα της σειράς των ε, ψηφοφοριών, των τροπολογιών, δεν σας δίνω το λόγο. Κύριε Συγήτρια, θέλετε να μιλήσετε για τη σειρά ψηφοφορίας των τροπολογιών. Καταρχήν, σε σχέση με το όσα είπατε, Madame la rapporteure. Pani Przewodnicząca, chciałam poruszyć dwa tematy przed głosowaniem. Proedra. ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Πριν ε, την ψηφορία έχουμε να δούμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με το εξή ότι οι συμβιβασμοί θα πρέπει να βασίζονται τουλάχιστον σε δύο τροπολογίες που κατατίθεται από δύο διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Δυστυχώ ο κατάλογος ε, των συμβιβαστικών τροπολογίων των σοσιαλιστών δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Πρόκειται για το ΑΑ, CCC, TDD, LL, MMM, DDD, EEE. Ε, ο συντονιστή τη ομάδα μα ε, σα έστειλε μια σχετική ενημέρωση, Πρόεδρε, προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά οι αντιδράσει μα δεν ελήφθησαν υπόψη από την Πρόεδρο. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τότε άτομο που είναι υπεύθυνο, που είναι αρμόδιο για τις τροπολογίες να μας απαντήσει για το θέμα αυτό και επίση θα ήθελα να μας εξηγηθεί από την νομική υπηρεσία γιατί πρέπει να δεκτούμε την απόφαση της Προέδρου σύμφωνα με την οποία η σειρά του των άρθρων 9 και 12 έχει τροποποιηθεί. Ε, ο συμβασμός ε, για το άρθρο 9 θα πρέπει να ψηφιστεί πριν από το συμβιβασμό Z2 των σοσιαλιστών, γιατί το κείμενο της Κομισιόν ε, εισαγάγεται ένα ανοιχτή λίστα μέτρων που θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην εισάγουν διακρίσεις και θα πρέπει να διαβιβάζονται πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ ο συμβασμός Z2 απλώς επιβάλλει το κατάλογο χωρίς κανένα όριο. Επομένως, ο συμβασμός LPL του Άλντε πηγαίνει πιο μακριά και πρέπει να ψηφιστεί πρώτα στο άρθρο 12, ο συμβασμός M1 Δια, διακόπτει την ομιλήτρια η Πρόεδρος, δεν έχετε πια το λόγο και θα σα απαντήσω για δύο θέματα. Για το πρώτο σημείο έλαβα ένα mail από τον Τζαμπαόρη, τον ε, συντονιστή σας και μου έγραψε στις 17 ε, Ιουνίου ε, του απάντησα μετά από λίγες, στις 10 η ώρα και εσείς ε, επίσης έχετε λάβει αυτή τη μελέτη, το απάντησα. Σας ευχαριστώ για το email σας ε, που θέτει κάποιες ανησυχίες ε, σε σχέση με κάποιες συμβαστικές τροπολογίες σοσιαλιστών. Έχω εξετάσει όλες τις τροπολογίες βάσει του ιστορικού κανονισμού δεν υπάρχει απέτηση συμβαστικέ τροπολογίες που καλύπτουν πάνω από μια τροπολογία ή να καλύπτουν τροπολογίες που να έχουν κατευθεί πάνω από μια ομάδα. Αντίθετα, σύμφωνα με τον κανόνα 161 παράγραφος 4, το παραδεκτό των συμβαστικών τροπολογιών πρέπει να αξιολογηθεί ανά περίπτωση ε, αξιολογώντας ε, την ε, φύση των συμβιβασμών. αυτών αυτό η προσέγγιση έχει ακολουθηθεί στο παρελθόν στην Επιτροπή μας. Το σημερινό έγγραφο δεν παρέχει πάντοτε πλήρες ενδείξεις σε σχέση με τις τροπολογίες που καλύπτονται που αντικαθιστούνται κατόπιν επαλήθευση μπορώ να σα επανεπιβεβαιώσω ότι καμία από αυτέ δεν έθεσε ανησυχίε καθώ ε, όλε ε, ε, αντικαθιστούν υφιστάμενε τροπολογίε. Ζήτησα όμω από την Γραμματεία να συμπεριλάβει στην τελική εκδοχή του εγγράφου και στον κατάλογο ψηφοριών όλε τι πληροφορίε, Υπό το φω των παρεπάνω αποφάσισα να θεωρήσω όλε τι συμβαστικέ τροπολογίε παραδεκτέ. Και θα διαβάσω τώρα για μια ακόμη ακόμη φορά το άρθρο 161 του ιστορικού κανονισμού και λέει σειρά των ψηφορίων των τροπολογιών έχουν προτεραιότητα στο κείμενο και το οποίο εφαρμόζονται. Αν ε, μία ή περισσότερε τροπολογίες που αμοιβαίως αποκλείονται ε, έχουν να κάνουν με το ίδιο τμήμα του κειμένου, τότε θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα η πρώτη και να απορριφθούν οι άλλες. Αν απορριφθεί, τότε ψηφίζουμε την ε, τροπολογία που ακολουθεί και αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την προτεραιότητα, τότε αποφασίζει ο πρόεδρο. Αν όλε οι τροπολογίε απορριφθούν, το αρχικό κείμενο θεωρείται ότι θετείται ε, εκτός και αν έχει ζητηθεί μηματική ψηφοφορία, ξεχωριστή ψηφοφορία μέσα στις εύλογες προθεσμίες. Λοιπόν, να ψηφίσουμε για το άρθρο 1, συμβασμό ΒΒ2 που έχει παρουσιαστεί από τρεις πολιτικές ομάδες. Υπέρ. Of opinion of tabling office. But you don't, this is the rule of the... Εγώ ζήτησα τη γνωμοδότηση του tabling office. Έχω το δικαίωμα αυτό, κυρία Πρόεδρε. Όχι, δεν απαιτείται εν, στην προκειμένη φάση. Έχω αυτό το δικαίωμα επιμένει η εισηγήτρια. Υπέρ κατά αποχές β ββ2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρασε. 21 ψήφοι υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. Β, Β1. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. 28 υπέρ, 18 κατά μηδέν αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 1, 1. Αλφα, αλφα, αλφα. Από δύο ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές. Παρακαλώ, επαλήθευση. Συμβαστική τροπολογία 3α. Παρακαλώ ψηφίσατε. Τέλος. 21 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 238 με μία προφορική τροπολογία, εφόσον δεν υπάρχει ένσταση κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Μα εκπίπτει αυτή. Άθρο 2, Παράγραφό 1. Συμβαστική τροπολογία ε2, ε, ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. η πρόεδρος. Συγγνώμη, έκανα κάποιο λάθος, διότι δεν εγκρίναμε την 3α, ααα δηλαδή, η οποία εκάλυπτε την 237. Για αυτό το λόγο πρέπει να ψηφίσουμε την ίδια την τροπολογία 237. Ψήφι υπέρ της 237 λοιπόν. Κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. Άρα έχουμε ψηφίσει τώρα την ε2 ε Συμβαστική ε1 από τρεις ομάδες. Υπέρ, κατά, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρασε. 28 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Προχωρούμε στο 2α, παράγραφο 16 της ε, Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 της ίδιας Επιτροπής. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομοίως. Άρθρο 2, παράγραφος 1, β. 18 της ε, Νομικής Επιτροπής υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται τι δω, αλλά ας επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Ψήφι 21 υπέρ, 25 κατά και όντως απερίφθη. Προχωρούμε τότε στις τροπολογίες 21 και 243 ταυτόσημες ψήφι υπέρ κατά. Υπέρ παρακαλώ, 21 και 243. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 και ζούρι 19. Ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 2-1. Τώρα, 234. 244 διορθώνει η πρόεδρος της κυρία Σόμεν Ρόιτεν και άλλων, καθώς και 242 Μπέκερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται αυτή. Καλώς, θέλετε επαληθευσή. Επαληθεύομαι λοιπόν την 244 και 242. Ψηφίσατε. Τέλος. ψήφι 21 υπέρ 24 κατά και μία αποχή. Όντως λοιπόν απερίφθη. 246 Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, με συγχωρείτε, ξέχασα τα 245. ...245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 της Επιτροπής ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 247 Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 3 Συμβαστική τροπολογία Α, Α1 από πέντε πολιτικές ομάδες, 4 μάλλον, υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. α, ΑΑ1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εφόσον ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Υπέρ 27, κατά 19. Η α 1 εγκρίνεται. Πηγαίνετε στη σελίδα 25 της λίστας παράγραφος 25 της νομικής επιτροπής στη σελίδα 25 της λίστας ψηφοφορίας. «24 του σοσιαλιστών, 25 των λαϊκών». Η φία 25 και για τη λίστα των ε, φιλελευθέρων. Λοιπόν, παράγραφος 25 της ε, Νομικής Επιτροπής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 3 μετά την παράγραφο 3. Ψηφίζουμε την συμβαστική ΠΠΠ δύο ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές θα επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρασε. 24 ψήφοι υπέρ, 20 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Μετά το άρθρο 3, συμβαστική τροπολογία ΒΒΒ, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, ας επαληθεύσουμε. Β, Β, Β. Ψηφίσατε, πέρασε. Ψήφι 23 υπέρ, 23 κατά. Άρα απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας. Ψηφίζουμε την 397 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται και αυτή, αλλά ας επαληθεύσουμε. 397. Ψηφίσατε. Τέλος. 21 ψήφοι υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. Μετά το 3β ψηφίζουμε την συμβαστική δέλτα δέλτα 2 τριών πολιτικών ομάδων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καλά, επαληθεύομαι. D, D2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. 23 υπέρ και 23 κατά. Άρα απορρίπτεται. Συμβαστική LLL, τρία λάμδα δηλαδή, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. συμβαστική τροπολογία Μετά από το άρθρο 3 ψηφίζουμε την συμβαστική δέλτα δέλτα 1 υπέρ. Κατά. Υπέρ D, DD1. Κατά. d DD1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρασε. 26 υπέρ. 20 κατά σαφώς εγκρίνεται. Μετά από το 3 γ ερχόμαστε στη συμβαστική τροπολογία D, 3 δέλτα δηλαδή υπέρ, κατά, αποχές, δεν εγκρίνεται. Συμβαστική 3 νι τριών πολιτικών ομάδων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ομοίως. Άρθρο 4. Συμβαστική σε δύο Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική σε ένα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 5. Συμβαστική Δέλτα 1. Συμβαστική τροπολογία Δέλτα 1. Υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Επαλήθευση για την D1. Ψηφίσατε, πέρας. 28 υπέρ, 17 κατά, σαφώς εγκρίνεται. Η Δέλτα 2 λοιπόν τότε εκπίπτει. Άρθρο 6. Πριν από το άρθρο 6, μετά το άρθρο 5, άρα μεταξύ των δύο, 5 και 6, η τροπολογία 461 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 6. Συμβαστική V2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική V1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται αυτή. Μετά το άθρο 6 η 484 494 μάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 7 W2 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. 21 ψήφοι υπέρ, 25 κατά, δεν εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν προχωρούμε στην W1 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Ψηφίσατε. πέρασε. «28 υπέρ 17 κατά». Έτσι λοιπόν εγκρίνεται καθαρά και αλλάζουμε σελίδα. Προχωρούμε στο άρθρο 8. Συμβαστική X2. X2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 6-1 υπέρ κατά αποχές αυτή εγκρίνεται. Αλλάζουμε σελίδα. Άθρο 9 συμβαστική Z2 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση Z2. Αρχίζει η ψηφοφορία. εφόσον ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. 27 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Και αλλάζουμε σελίδα. Σελίδες μάλλον. 60 λοιπόν, σελίδα 60. Και μάλιστα 62. Στο τέλος του άθενια, το, 600, το πρωί 615 υπέρ 615 μετά το άθενια. υπέρ κατά αποχές επαλήθευση αν και νομίζω ότι απορρίπτεται Ψηφίσατε πέρας. 20 υπέρ, 25 κατά. Όντως λοιπόν απερίφθη και ε, μια αποχή. 613 της Αντιπροέδρου Χίρς υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε. Πέρας για την 613 διορθώνει η πρόεδρος. Έκλεισε τώρα, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Υπέρ 21 ψήφι κατά 22 και 3 αποχές, άρα απορρίπτεται. Τώρα, τροπολογία 616 και προτιμώ να ψηφίσουμε ευθύς αμέσως ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. 21 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. Και καμία αποχή, άρα απορρίπτεται. Άρα μπορούμε να θέσουμε σε ψηφοφορία την υπαριθμό 614 του κ. Χέντελ υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. Άρθρο 10. Τροπολογία σε, σε 1. Υπέρ. Κατά αποχές. Επαλήθευση. σε, σε ένα. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Τέλος. Ψήφι 28 υπέρ, 18 κατά, άρα εγκρίνεται. Προχωρούμε. προς το τέλος των σελίδων 60 κλπ. Και μετά το άρθρο 10, συμβαστική τροπολογία 3ε, ε, ε, ε δηλαδή. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 644 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και αυτή. 647 της κυρίας Σρόιντερ και Κρυσιάς Υπέρ. Α, με συγχωρείτε αυτή εκπίπτει. Αν όχι, πάλι με συγχωρείτε, δεν εκπίπτει λέει η πρόεδρος. Κατά το έλεγα. Άρα, 647 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται και αυτή. Καλά, επαλήθευση λοιπόν για την 647. Tout le monde a pu voter. υπέρ κατά 25, άρα δεν εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την διακό. λέει πρόεδρος και διακόπτη. Ψηφίζουμε τη 220 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε. Επαληθεύουμε για τη 220. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 20 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. Στο άρθρο 11 ψηφίζουμε το συμβασμό FF2 υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σκόπιμο θα ήταν να υπαλληθεύσουμε. Πέρας. 21 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τροπολογία συμβασμού FF1. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά καλύτερα. FF1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 28 υπέρ, 18 κατά. Άρα εγκρίνεται. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στο άρθρο 12, άρθρο 12, Έχουμε 7 τροπολογίες διαγραφής. Εάν τις ψηφίσουμε, δεν ψηφίζουμε την τροπολογία συμβασμού. Το, καταλα... το κατανοείτε αυτό. Ποιος είναι υπέρ της διαγραφής του άρθρου 12. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 16 υπέρ 31 κατά, άρα απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το συμβασμό MM2, αρχίζει η ψηφοφορία, λέει η πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 25 υπέρ, 21 κατά, μία αποχή, άρα εγκρίνεται. Euh, Στον κατάλογο βλέπουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο άρθρο 13, σελίδα 84. Άρθρο 13, εφόσον έχει διαγραφεί το 12. σελίδα 84 στο ελληνικό κείμενο. Άρθρο 13, GG2, υπέρ. Άρθρο 13. Συμβιβασμός GG2, υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. GG2. Επαληθεύουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 26 κατά. Πράγματι απορρίπτεται. GG1 τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, αλλά θα επαληθεύσουμε παρόλα αυτά. Le vote clos. Πέρας. 28 υπέρ, 18 κατά. Πράγματι εγκρίνεται. Άρθρο 14 τωρα συμβιβασμος Συνδυασμός HH2. Δύο ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Συμβασμός HH1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά το άρθρο 14, παράγραφος 45 ε, της Νομικής Επιτροπής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 15. Ψηφίζουμε δύο πανομοιώτες JJ1 και JJ2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Στο άρθρο 16 δύο πανομοιότυπες ΚΚ1 και ΚΚ2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Μετά το άρθρο 16, λέει πρόεδρος και διακόπτη, Ωραία. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε το άρθρο 16 λοιπόν. Τις δύο τροπολογίες συμβασμού. ΚΚ1 και ΚΚ2. Ζητώ συγγνώμη για το κακό ήχον των τροπολογιών. Τώρα ψήφισαν όλοι. Πέρας. 42 έναντι 5. Άρα εγκρίνονται. Ε, και σας ευχαριστώ για την επαλήθευση χαλαρώσαμε λιγάκι. Μετά το άρθρο 16 έχουμε δύο πανομοιότυπες. Θέλετε να τις επαληθεύσουμε πάρα αυτά LL1 και LL2 που είναι παρομοιότυπες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το άρθρο 17, 804, Σρέτερ και Τουρνέν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά το άρθρο 19 ψηφίζουμε την 825 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 805 Τόμας Χέντελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 806 Τόμας Χέντελ υπέρ κατά αποχές ε, ας ελέγξουμε. 806 επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 22 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. 807 του ιδίου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 808 του ιδίου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 809 του ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 810 του ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 811 του ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 18. Συμβεβασμός Y1 υπέρ. Κατά Αποχές ε, εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε όμως καλύτερα. Συμβασμός Y1. Y1. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Η 20 είναι υπέρ, 15 κατά, 3 αποχές. Γυρνάμε σελίδα. Μετά το άρθρο 19, τροπολογία 820, 826, Σρέτερ και Τουρούνεν, όπου υπάρχει και μία προφορική. Δεν αντιτίθεται κάποιος, ψηφίζουμε την 826 όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 827 των ιδίων για το άρθρο 20 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 828 των ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στο άρθρο 21 παράγραφος 1 τροπολογία 830. Μάλλον στον τίτλο, στον τίτλο 829 Τόμας Χέντελ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, τροπολογία 830, Τόμας Χέντελ, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 831, Μπουλάν Μορέν Σαρτιέ, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 832, Χάρκιν, υπέρ. Κατά, αποχές, Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. Ελέγχουμε για την 832. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 26 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Έχοντας υπόψη 59 Σρέτερ και Τουρούνεν υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 60 και 61 πανομοιότυπες ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Μετά το έχοντας υπόψη 1, 64 του Ρούνιν και Σρέτερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, έλεγχος, τροπολογία 64. Μάλλον έκανα λάθος για μία φορά. Πέρας. 26 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Σαφώς. Άρα εκπίπτει η 62 και 63. Ε, έχοντας υπόψη και εδώ ψηφίζουμε την τροπολογία 65. Χιούς και άλλοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στέχοντας υπόψη 2, 1 τις ε, και ΙΜΚΟ πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε, ελέγχουμε για την υπαριθμόν 1. Πέρας 25 υπέρ, 21 κατά και μία αποχή, άρα εγκρίνονται. Μετά το έχοντας υπόψη 2, 68 Τόμας Χέντελ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά το 2α, ΙΜΚΟ 2 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 69 ε, Χέντελ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 70 Σρέντερ Τουρούνεν υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 71 των ιδίων υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται στο έχοντας υπόψη 3, τροπολογία 73, Σρέτερ του Ρούνεν, η ίδια με την παράγραφο 2, με την ΙΜΚΟ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 72 του Τόμας Χέντελ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 74. Ποιους και άλλων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη 3.76 Σρέτερ του Ρούνεν και παράγραφος 4 της ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 Στίβεν Χιούς και άλλων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 77 Λούντβιξον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 78 Στίβεν Χιούς και άλλων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά το, την αιτιολογική σκέψη 3, ΙΜΚΟ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη 3, 79 Στίβεν Χιούς και άλλων υπέρ Θέλετε να ελέγξουμε. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά το είναι αιτιολογική σκέψη 4 τροπολογία 85 Σρέντερ και του Ρούνεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 84 Νάντια Χίρς με μια προφορική προοπτική της ιδίας Κανείς δεν αντιτίθεται, άρα ψηφίζουμε την τροπολογία 84 όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 4. συμβασμο 1 1-2 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε έν, έν, 1 με συγχωρείτε λέει η προεδρος NN1. Επαλήθευση. Πέρας. Ψηφίσατε όλοι ελπίζω. 26 υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη 4, 86 μεταξύ 7 ΙΜΚΟ και 2 της Γιούρη που είναι πανομοιότυπες. Ψηφίζουμε, η συγγήτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Στο 5, τροπολογία 87, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 8 της ΙΜΚΟ Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το 5, παράγραφος 9 της ΙΜΚΟ Κατά αποχές απορρίπτεται στην αιτιολογική σκέψη. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε. Λοιπόν, ΙΜΚΟ 9, ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 26 υπέρ 17 κατά. Είχετε απόλυτο δίκιο με τρεις αποχές. Εγκρίνε. Στην αιτιολογική σκέψη 6 FFF 2 ομάδων υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Προχωράμε. Μετά την 6 στην παράγραφο 3, την παράγραφο 3 της Γιούρη. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 της εισηγήτριας και άλλων υπέρ. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. 90 λέει η πρόεδρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 91. Τόμας Χέντελ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 92. Σρέτερ και Τουρούνεν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά το 7 παραγραφός 11. Ήμκο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στο 8 συμβασμός PP2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός PP1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε τον συμβιβασμό, την πρωτη συμβασμο συμβιβασμού PP1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 25 υπέρ, 21 κατά, μία αποχή Πράγματι εγκρίνεται. Μετά το 8, 98 Τόμας Μάν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το 9 ε, συμβασμός τριπλό G υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά 89. Ψηφίστε παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αμόνο. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε παληθεύσουμε καλύτερα. Ψηφίσουμε την 100, επαληθεύουμε. Vote Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 18 υπέρ, 25 κατά, 3 αποχές απορρίπτεται μετά το 9, τροπολογία 101 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Στο 10 Τροπολογία συμβιβασμού QQ1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. QQ1. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 25 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. Τις δεν εκτιμώντα 10, πάμε στο συνδεσμό RR1 υπέρ. Υπέρ. Για το συνδεσμό RR1. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Μετά το εκτιμώντας 10 πάμε στην τροπολογία 112 και η τροπολογία 113 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά Αποχές. απορρίπτονται. Τιμώντας 11 συνδεσμός ο μικρονό μικρον 1 υπέρ κατά Αποχές. εγκρίνεται. Μετά πάμε στην τροπολογία 117, στην Βενχιούς. Υπέρ, κατά, αποχές. Να επαληθεύσουμε για την 117. Άρχεται ψηφοφορία. Έχουμε έναν υπεράριθμο σοσιαλιστή και ο Μπούλμαν μπορεί να φύγετε, Συμφώνησαν στους σοσιαλιστές για το θα ψηφίσει. Πέρασε. 21 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας 12, συμβασμός SS, υπέρ, κατά, αποχές. Να επαληθεύσουμε το συμβασμό αυτό, SS. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι έχουμε έναν υπεράριθμο σοσιαλιστή. Ωραία, πέρας. 29 υπέρ, 14 κατά, 3 εποχές. Γκρίνεται. Μετά, τροπολογία 124, το μασμάν υπέρ. Κατά, εποχές, γκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε, εγώ έχω την εντύπωση ότι ευρέως υιοθετείτε. Παράγραφος 4. Ε, Επιτροπή Γιούρι, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 16 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Έχουμε τώρα το συμβασμό TT1 για το 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Να επαληθεύσουμε το TT1 αλλά Ξέρετε, μερικές φορές δεν σηκώνετε τα χέρια. το όλοι πέρας. 24 υπέρ, 22 κατά. Έχετε δίκιο, να κρίνετε. Ψηφίζουμε με τα δοκτήματος 14, τις τροπολογίες 125, Παράγραφος 18 ΙΜΚΟ με έτοιμα τμηματικής ψηφοφορίας. Ε, λοιπόν, πρώτο τμήμα του κειμένου χωρίς τον όρο φύσιλ, Την 135 και 18 ΙΜΚΟ υπέρ. Ποιος είναι υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά εποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ για την προσθήκη του φύσιλ, υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουν. Ψήφισατε όλοι, πέρας. «23 υπέρ, 23 κατά». Δεν εγκρίνεται. Περνάμε στο κτήμα 15, συμπεσμος uu UU1. δυνατόν να δουλέψουμε έτσι. Λοιπόν, συμβεσμός συνδεσμός ένα. υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται να το επαληθεύσουμε όμως. Πέρας. 29 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Λοιπόν, έχουμε την τροπολογία 137 τώρα, Σρέτερ του Ρούνεν, παράγραφος 19, τη ΣΥΜΚΟ, ταυτόσημες, υπέρ. Κατά, εποχές, απορρίπτονται. Εκτιμώντας 16, συνδεσμός VV1, υπέρ. Κατά, εποχές, να επαληθεύσουμε το συμβασμό VV1. in the middle of the vote in the, in, in the tribune, it's not possible. Donc le vote est clos. Πέρασε ψηφορίας. 22 υπέρ, 24 κατά, δεν εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το συμβασμό VV2. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 24 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Μετά το εκτιμώντας 16 περνάμε στην τροπολογία 150 και την παράγραφο 21 της Συνικού υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε παλήθευση. Εκτιμώντας 17, συμβασμός WW1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συνδεσμός Λοιπόν, επαλήθευση για το WW1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 28 υπέρ, 19 κατά, έχετε δίκιο. Εγκρίνεται με σαφήνεια, έτσι λοιπόν. Περάμε στην τροπολογία 153 αναδιαχείριση, υπέρ. Περ. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 114. Χιούς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτει. 155 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα χωρίς τον όρο blacklist. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει το πρώτο τμήμα. Πάμε στον 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 157 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα χωρίς τους όρους ασφαράς possible υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Ψηφίζουμε την παράγραφο 22 της Πεσίνικο, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 158 το Μασμάν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 20, τροπολογία 159. Εδώ ζητείται διαγραφή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 160 του Ρούνεν και Σρέτερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 συγγνώμη 10 της εισηγήτρης υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε για τη 10 άρχεται ψηφορία 25 υπέρ, 19 κατά, 4 εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 τη υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Είμαστε 22, τροπολογία 161 του μασμάνι υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση για την 161. Ψήφισατε όλοι, πέρας. 26 υπέρ. 21 κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8 της Επιτροπής των Καθημάτων Καταπίπτη, εκτιμώντας 23, ψηφίζουμε την τροπολογία 12 της συνήθειας. Τι έχει γίνει με το 2 γιατί έχει περάσει και ώρα από τότε που το ψηφίσαμε. Και για το άρθρο 11. Καταπίπτει λοιπόν η τροπολογία αυτή. Λοιπόν, καταπίπτει το είχε καταπέσει το 2, μπορούμε να το ψηφίσουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε τροπολογία 12, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε για την τροπολογία 12 της εισηγήτριας. Ψήφισατε όλοι, πέρας. 25 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. Επομένω, τροπολογίε 163 και παραγράφους 24 τούτων. και 162 και 164 και πάμε στο κτήματος 24 όπου έχουμε 7 τροπολογίες που ζητούν τη διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ της διαγραφής του κτήματος 24, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφορίας. 25 υπέρ. 22 κατά. Εγκρίνεται. Δεν ε, υπάρχει πλέον συμβιβασμό λοιπόν. Πάμε στο κτήμα 25. Και εδώ Έχουμε δύο τροπολογίες που συμβαστικές που ζητούν τη διαγραφή. Και μετράει η πρόεδρος. 11 τροπολογίες που ζητούν τη διαγραφή. Του εκτιμώντας 25, δεν είμαι και σίγουρη ότι θα παραμείνει. Ψηφίζουμε υπέρ. Υπέρ της διαγραφής του 25. Κατά αποχές θέλετε παλήθευση Υιοθετείτε λοιπόν. Με το 25 έχουμε την τροπολογία Χέντελ 188 υπέρ. Και το πίπτον, γιατί διαγράψετε το εκτιμώντας. 188 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτει. Κομμάτις 26. Συμβασμός Ι1 και Ι2 καθώς και 10 τροπολογίες 12 συνολικά προτείνουν τη διαγραφή του εκτιμώντας 26. Ποιος είναι υπέρ της διαγραφής του 26 κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά λοιπόν το εκτιμώντας 26 πάμε στην τροπολογία 199 υπέρ. Κατά αποχές απαραίτητα. Μετά το εκτιμώντας αυτό πάμε στην τροπολογία 200 υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε για την τροπολογία 200. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. 18 υπέρ, 22 κατά. 7 αποχές. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας 27. Τροπολογία της εισηγήτριας. 16. Ζητά τη διαγραφή υπέρ. Κατά. Αποχέες. απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο 28. Συγγνώμη, να επαληθεύσουμε για τη 16 της εισηγήτρης. Ψηφίσατε όλοι. Έχουμε υπεράριθμο στο ΕΛΚ. Κύριε Ωρή, πρέπει να διαλέξετε. Πέρας. 25 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Επομένω, καταπέπτουν οι ακόλουθε τροπολογίε και πάμε στην τροπολογία 17. Ζητάει η συγκεκριτή διαγραφή του εκτιμώντα 28 υπέρ. Εντάξει, αν ε, εγκριθεί 17 θα μπορούμε να ψηφίσουμε για το συμβασμό και καθώς το ΕΛΚΑ έχει εκπονήσει συμβασμούς θέτω σε ψηφορία τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επελθεύσουμε. Άρχεται η ψηφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 18 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. Επομένω ψηφίζουμε το συμβασμό YY1 και YY2 που είναι ταυτόσιμοι. Υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε για τους συμβασμούς YY1 και 2. Άρχεται η ψηφορία, ψηφίστε τα όλοι πέρας. 42 πέρ. 5 κατά, καμία εποχή. Εγκρίνονται. Μετά λοιπόν από το 28 φτάνουμε στο τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτήματος 29, δύο τροπολογίες ταυτόσιμες, 204 και μκο 30 υπέρ. Κατά εποχές Δεν σηκώνετε τα χέρια για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για αυτές τις δύο. Την 24 και την 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 25 υπέρ, 18 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται. Κτιμώντας 30, τροπολογία 19 της 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 31, 207 του Τόμας Μαν. Υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε για τη 207. Άρχεται η ψηφορία, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 21 υπέρ. 24 κατά. Και έχασε ο Λυπάμαι. Επομένω, καταπίπτει και φτάνουμε. Στο τη 33, τροπολογία 213 υπέρ. 213 υπέρ κατά για τη 213 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Σφίζουμε τη 214 του Ρουνού και Σρέντερ υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Μετά Περνάμε στην τροπολογία 215, στα υπέρ, κατά, ποιες απορρίπτεται. Εκτιμώντας 34, τροπολογία 216, το μασμάν υπέρ, κατά, ποιες απορρίπτεται. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου της έκθεσης ηλεκτρονικά. έρχεται η ψηφοφορία. Υπεράριθμη το ΕΛΚ. Πέρς. 20 υπέρ, 18 κατά, 6 εποχέ. Λοιπόν, ψηφίσουμε την νομοθετική πρόταση έτσι όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 22 υπέρ, 18 κατά, 6 εποχές. Τώρα θα ψηφίσουμε την εντολή είναι ξεκαθαρά όλα ή θέλετε διακοπή της σας κάποιοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει κυρία Τώρα θα ψηφίσουμε την εντολή. Δεν θα ήταν καλύτερα πρώτα να πάμε στην Ολομέλεια. Χθε έτσι κρίναμε στην ομάδα του Λαϊκού Κόμματος. Πρώτα να πάμε στην Ολομέλεια. Και εγώ προσωπικά το βρίσκω αυτό καλύτερο. Ας διαθέσουμε ένα λεπτό στο σημαντικό αυτό στο στάδιο της συζητήσεως, δηλαδή αν θα προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις ή όχι. Σας παρακαλώ, ησυχία. Δυνάμει του άρθρου 66 του κανονισμού μας, αν θέλουμε να ανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις στην βάση της εντολής όπως καθορίστηκε, μας χρειάζονται 25 ψήφοι υπέρ της έναρξης των διαπραγματεύσεων. Προτείνω δύο λύσεις. Εάν κάποιες πολιτικές ομάδες επιθυμούν να διακοπεί η συνεδρίαση για να εξετάσουν τη θέση τους, ευχαρίστω να τους το δώσω. Η άλλη επιλογή είναι, που σας προτείνω επίσης, να επιτρέψουμε σε κάθε ομάδα να τοποθετηθεί για την θέση που επιθυμεί να λάβει για την εντολή, για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Τρίτη λύση είναι συνδυασμός των δύο. Δηλαδή να γίνει μια σύντομη διακοπή της συνεδριάσεως και μετά κάθε ομάδα να λάβει τον λόγο για να εξηγήσει την θέση της σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Αν έχω καταλάβει καλά, είναι σύμφωνο το Λαϊκό Κόμμα. Ας διακόψουμε για πέντε λεπτά τη συνεδρίαση. Bien. Si tout le monde veut bien reprendre. Η πρόεδρος, παρακαλώ καθίστε πάλι. Καλά λοιπόν. Ο κύριος Όρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ψηφοφορία δεν έγινε όπως αναμέναμε ή δεν απέδωσε αυτά που αναμέναμε. Εμείς πάντως είμαστε υπέρ της χορηγήσεως της εντολής, δοθέντος ότι είναι παρόλα αυτά επαρκής η βάση. Ο κύριος Θέρκας, ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική στιγμή της θητείας μας και πιθανότητα με το νομοθέτημα που αναμένουν ευρύ τομείς της ευρωπαϊκής κοινωνίας και ενηλικεί ότι αυτή τη στιγμή έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση όπου και η δική μας επιτροπή είναι ιδιαίτερα διχασμένη, βάθος διχασμένη, δεν έχει αναζητήθει μια συμβιβαστική θέση αλλά μια θέση ιδιαίτερα αποσχεστική και έτσι τελικά έχουμε ένα διαιρεμένο κοινοβούλιο και δεν επιτρέπεται να έχουμε μια λογική διαπραγμάτευση εδώ γιατί τελικά βλέπουμε να υπάρχουν και αντιφατικά επιχειρήματα και αποφάσεις. Έτσι λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση το να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο θα είναι σαν να μπαίνουμε στις διαπραγματεύσεις αποδυναμωμένοι και συγχυσμένοι και έτσι ε, τελικά θα είναι σαν να ε, μπαίνουμε ιτημένοι στη διαδικασία αυτή και να μην κάνουμε καμία προσπάθεια για να λύσουμε ένα πρόβλημα για εκατομμύρια εργαζομένους ε, και σε πολλές χώρες που δεν θα έχουν ασφάλεια δικαίου στις εργασίες τους σχέσεις όταν εργάζονται σε άλλη χώρα. Έτσι λοιπόν εγώ νομίζω ότι αν κάποιος ξεχάσει τις ε, ε πολιτικές κομματικές θέσεις ε, θα ήταν καλό να προσπαθήσουμε να βρούμε συμφωνία μεταξύ μας πριν από την Ολομέλεια για να έχουμε μία ε, πιο χρήσιμη θέση και πιο συμβιβαστική έτσι ώστε να μπορούμε να λάβουμε και μία βελτιωμένη θέση απέναντι στο Συμβούλιο. Εμεί ζητάμε, λοιπόν, η ομάδα μου ζητάει να μην ψηφίσουμε αυτή την εντολή, γιατί μα αποδυναμώνει και μα διχάσει και να προσπαθήσουμε στην Ολομέλεια να ενωθούμε και να ενδυναμωθούμε. Κύριε Χίρση, για του φιλελεύθερου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εμείς διαβουλευθήκαμε, είδαμε ότι πολλές από τις θέσεις που ψηφίστηκαν ήταν ορθές και προτιμούμε και εμείς να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις και επομένως να δοθεί σήμερα η εντολή στην διαπραγματευτική ομάδα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να δούμε και τι απόσταση έχουμε εν τέλει και από το Συμβούλιο. Τζιν από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Και εμείς θεωρούμε ότι οι σημερινές ψηφοφορίες κινήθηκαν προς θετική κατεύθυνση. Έτσι στηρίζουμε και εμείς την χορήγηση της εθελοντής ε, ε, διαπραγματικής στολής. Ε, εκ μέρους των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών παρετείται. Τώρα για την ενωτική αριστερά μιλεί ο κύριος Χέντελ. Εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι επαρκές το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις και είμαστε κατά της χορήγησης της σχετικής εντολής. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος του Α, με συγχωρείτε. Υπάρχει. Ο κ. Στερό. Καλά λοιπόν, μετά την απάντησή σας θα θέσω... να τι είπε, δεν καταλάβαμε. Λένε ορισμένοι βουλευτές, ούτε και οι διερμηνείς κατάλαβαν, δεν πρόλαβαν να ακούσουν τίποτα. Κύριε Τερό, μπορείτε να επανατοποθετηθείτε σας παρακαλώ. Να δοθεί η διαπραγματευτική εντολή. Α, θαυμάσια, το λέει και στα αγγλικά. We support. J'ouvre donc le vote. Άρα, αρχίζει η ψηφοφορία για την χορήγηση της διαπραγματευτικής εντολής στη βάση των ψηφοφοριών που διεξήχθησαν σήμερα στην Επιτροπή. Υπενθυμίζω ότι χρειάζονται 25, 25 ψήφοι υπέρ. Ψηφίσατε όλες και όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 30 ψήφοι υπέρ, 17 κατά. Επομένως, χορηγείται η εντολή. Παρακαλώ, δεν τελειώσαμε ακόμα τις ψηφοφορίες. Η εισηγήτρια ζήτη να λάβει το λόγο, ωστόσο. Τη δίνω το λόγο. Κύριε εισηγήτρια, παραμείνετε καθιστή, παρακαλώ. Παραμείνετε καθιστή. Έχουμε ακόμα δύο ψηφοφορίες. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να είστε σχετικά σύντομοι, όλα αυτά σας δίνω ευχαρίστω στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους ε, βουλευτές, βοηθούς, ε, τη γραμματεία, όλους ε, όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτό το έγγραφο για την προστασία των εργαζαμένων και τους αποσπασμένους. Ευχαριστούμε και τη Γραμματεία γιατί μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη ψηφοφορία που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Σημείο 36. Έκθεση Χέντελ για τις διασυνοριακές συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον διεθνικό κοινωνικό διάλογο. Πριν από την παράγραφο 1, 42. Όλα Λούντβικσον υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 1. Συμβασμός C υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. S'il vous plaît, on est au milieu du vote. Σας παρακαλώ ψηφίζουμε. Θα ήθελα λίγη ησυχία στην αίθουσα. Παράγραφος 2. Ντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2 τροπολογία 55. Λούντβικσον υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56. Ζαν Πιεροντή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται για τους υπότιτλους, υποκεφάλαια 57 κορνέλησαν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58 των ιδίων υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Ελέγχουμε την 61. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 22 υπέρ, 23 κατά, δεν εγκρίνεται, 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 63 υπέρ, κατά, αποχές, 63 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε, 63 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Πέρας. 20 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στον υπότιτλο 1, μία διαγραφή 65 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68. Θέλετε να ελέγξουμε 67. Ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 19 υπέρ, 25 κατά απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 κοτσολίνο αποσύρθηκε, άρα ψηφίζουμε την 70 εσάγια υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Συμβασμός ε τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν το συμβασμό ε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 21 υπέρ, 23 κατά. Άρα πράγματι απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε την 72 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν ψηφίζετε πλέον. 72. Παρακαλώ ψηφίστε υπέρ. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τελικά. Πέρας. 22 υπέρ 21 κατά εγκρίνεται. Οι άλλες εκδίπτουν. Παράγραφος 5.76 αποσύρθηκε. Άρα ψηφίζουμε το συμβασμό F τριών πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρο F. Πέρας. 35 υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Τρεις ε, τροπολογίες ε, διαγραφής 82, 83, 84 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. «89 υπέρ». 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 ε, Λούτβικσον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 κλειβέτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 Λούτβικσον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Τρεις, ε, τροπολο... Τέσσερις τροπολογίες διαγραφής τις ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές ε, ελέγχουμε γιατί δεν ψηφίζεται πλέον, δεν συμμετέχετε. Υπέρ της διαγραφής της παραγράφου 7. Αρχίζει η ψηφοφορία πέρας Ισοψηφία 20-20 απορρίπτονται. Ψηφίζουμε λοιπόν την 97 τσάμπα όρη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8, 99 Μπέκερ για διαγραφή. Όχι, πριν πρέπει να ψηφίσουμε την 98 του εισηγητή. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 899 Πέκερ για διαγραφή ΠΕΡ. κατά αποχές ελέγχουμε. 99 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. Ισοψηφία 21-21 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τον συμβασμό H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 9, τέσσερις ε, τροπολογίες διαγραφής της παραγράφου 9. Υπέρ της διαγραφής παραγράφου 9, κατά αποχές επαληθεύουμε. Για τη διαγραφή της 9. Ψήφισατε όλοι πέρας 22 εναντί 20, άρα εγκρίνονται. Καταπίπτει ο συμβασμός παράγραφος 10 με 5 διαγραφή, τροπολογίες διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ της διαγραφής παράγραφου 10, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται η διαγραφή της παραγραφού 10, ελέγχουμε. Ψήφισατε όλοι πέρας. 22 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 122, εσάγια υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος, 122, ελέγχουμε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 15 υπέρ 22 κατά 5 αποχές πράγματι απορρίπτεται. Τροπολογία 123 Λούδβιξον υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 124 Κορνέλισεν Σρέντερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στην παράγραφο 11 η 125 για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το συμβασμό Κ. Τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με την παράγραφο 12 τρεις τροπολογίες διαγραφής υπέρ της διαγραφής παραγράφου 12 κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη διαγραφή της παραγράφου 12. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. ισοψηφία, μάλλον όχι, δύο υπέρ, 20 κατά, άρα πράγματι εγκρίνεται. Μετά παραγραφό 12, 13, 137, Λούντβιξον υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 138 κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 Λούτβικσον. επαλήθευση 138 Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 36 υπέρ, 6 κατά. Κάτι συνέβη, κάτι συνέβη, δεν μπορεί. Εγκρίνεται. Ε, με μεγάλη πλειοψηφία. 139 Λούδιξον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140 του ιδίου υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Έλεγχος 140. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ. 16 κατά. 5 αποχές. Έγκρινεται 141 του ιδίου υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτε 142 του ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 του ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά την παράγραφο 13 συμβασμός M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά παράγραφο 13 14 144 Νάτια και άλλων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στα έχοντας υπόψη 1 Λούδικσον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2 Λούδικσον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 3 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 5 Κορνέλισεν υπέρ. Σρέτερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17, τρεις ε, τροπολογίες διαγραφής. Ποιος είναι υπέρ της διαγραφής του 17, υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε για τη διαγραφή του έχοντας υπόψη 17. Ψήφισα το όλοι πέρας. 20 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την 11 του Λούδβιξον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 του ιδίου. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Έλεγχος 11. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 21 υπέρ, 16 κατά, 4 αποχές εγκρίνεται. 12 του ιδίου υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 του ιδίου υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται στο β στην αιτιολογική σκέψη Β ψηφίζουμε την 19 στο Β, 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 19. Ψηφίζουμε. Έλεγχος. Ε, ο εισηγητής είναι κατά. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 19 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Α, καταπίπτει 20. Με συγχωρείτε, 21 και 21 στο C, τροπολογίες 22 και 23 υπέρ, για τη διαγραφή, υπέρ της διαγραφής δηλαδή. Κατά αποχές εγκρίνονται. Στο Δέλτα 26 χείρς και άλλων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το Δέλτα 27 Λούντβιξον υπέρ. Κατά αποχές απόρριπτα 28 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται στο ε τροπολογία 29 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβατεί 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά το ε, τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Μετά το ε, 32 Κορνέλισεν Σρέτερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στο F33 Σαριεσάια υπέρ κατά αποχές ε, δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε 33. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας 33. Όχι, ψηφίζουμε την 33. Σάρι 33. Ο εισηγητής είναι κατά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 21 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την 34 Κορνέλησεν. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το G, συμβασμός Β. Ο συμβασμός αυτός έχει αποσυρθεί. Άρα ψηφίζουμε την 35 υπέρ. 35. Ψηφίζουμε. Ο συγκρίτης είναι κατά. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Το C της ΦΑΜ εκπίπτει, άρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να ελέγξουμε τη 40, θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, ωραία, ελέγχουμε τη 40. Ψηφίζουμε, ελέγχουμε για την 40, ψηφίσατε όλοι. 21 υπέρ, 20 κατά. Πράγματι λοιπόν εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 31 6 κατά, 3 αποχές. Να συγχαρούμε τον εισηγητή μας. Σα προτείνω να συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρία τη επιτροπή μα ε, τα θέματα που μας απομένουν στην ημερησία διάταξη. Τα τρία αυτά τα βάλουμε για την επόμενη φορά. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ και του διερμηνείς. Και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη συνεδρίασή μας στις 8 Ιουλίου.